έχω να σας κάνω την ε, λυπηρή ε, ανακοίνωση ότι ο Κίνιος Πέισλε την προηγούμενη Παρασκευή πέθανε σε ηλικία 88 ε, ετών. Ήταν επί μακράων βουλευτής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο τέλος της θητείας του εδώ πέρα διατέλεσε και υπουργό στην Ιρλανδία. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι να σας ενημερώσω ότι πολλοί συνάδελφοι μου επέστησαν την προσοχή το εξής σήμερα λαμβάνουμε τώρα, δηλαδή που σας μιλάω, λαμβάνουμε νέες δραματικές ειδήσει για ναυάγια, δραματικά ναυάγια. 500 οι ε, θάνατοι εικάζονται στην Μεσόγειο. 36 ενδεχομένως να σωθούν, αλλά ε, περίπου 200 είναι τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τη, ε, Έξω από τις ακτές της Μάλτας λοιπόν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 500 άτομα. Νομίζω ότι έχουμε ηθικό χρέος να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας κυρίες και κύριοι για να προλάβουμε στο μέλλον περαιτέρω τέτοιες ανθρωπιστικές καταστροφές τις οποίες δεν μπορούμε πραγματικά να επιτρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα σας ανακοίνωσα και θα ήθελα εδώ να το επαναλάβω ότι αύριο, λίγο πριν την ψηφοφορία, εδώ θα γίνει μία μαγνητοσκόπηση, α, συγγνώμη, όχι αύριο, την Τετάρτη, πριν την ψηφοφορία, λοιπόν, 360 μοιρών. Όλα, λοιπόν, τα μέλη θα καταγραφούν με μια τέτοια κάμερα περιστροφική. Ξέρετε, λοιπόν, έχουμε κάνει μια τέτοια μαγνητοσκόπηση 360 μοιρών. Παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ πέρα γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές δυνατότητες για να ελέγξουμε και να δούμε πού βρίσκεστε ως βουλευτές εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας και οι επισκέπτες μας θα μπορούν λοιπόν να παρακολουθήσουν και συνάδελφοι θα το συζητήσω και με τον κύριο Ρόιλ το θέμα αυτό. στι 12 λοιπόν ε, το μεσημέρι την Τετάρτη μαγνητοσκόπηση 360 μοίρων. Τα πρακτικά τη συνεδρία τη 17, η Ιουλίου έχουν διατεθεί στου βουλευτέ, Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Άρα λοιπόν εγκρίνονται τα πρακτικά. Κυρίε και κύριοι, έχω μια σειρά ανακοινώσεων να σα κάνω. καταρχά. οι αρμόδιες, οι αρμόδιες ισπανικές αρχές